να με τους εταίρους μας ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της Ερυθρέας. Το διάλογο αυτό λοιπόν, αλλά και δημόσια, με τις ανησυχίες μας σχετικά με τις παραβιάσεις της Ερυθρέας που δεν τηρεί και δεν προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα. Χρειάζονται συγκεκριμένες χειρονομίες ελευθέρωση των κρατουμένων που βρίσκονται στο Κομμουνικάντο από το 2001 για παράδειγμα και κυρίως τον κύριο Νταβίτισαν και άλλους Ερυθρέους πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης τις ανησυχίες αυτές τη θέτει και σε διάφορα φόρα στο Συμβούλιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, για παράδειγμα, όπου ζητάμε συνεργασία με τον ειδικό απεσταλμένο του ΟΗΕ και με την Ερευνητική Επιτροπή για την Ερυθρέα, προκειμένου να μπορέσουν να πάνε στην Ερυθρέα. Νομίζω ότι η καλύτερη λύση για διάφορους λόγους είναι να συνεχίζουμε τις επαφές μας με την Ερυθρέα. Πρώτα απ' όλα γιατί η σχέση αυτή βοηθάει να υπάρχουν ευκαιρίες για σημαντικές αλλαγές και πρόοδο. Επιμένουμε επίσης ότι πρέπει να έρθει στις διεθνείς προδιαγραφές η Ερυθρέα. Δεύτερον, επειδή μόνο έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον πληθυσμό επιτόπου και να βελτιώσουμε έτσι τις συνθήκες ζωής του. Και τέλος, επειδή με την σχέση αυτή ενισχύεται η σταθερότητα και στη χώρα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει κάποια πρόοδος τελευταία. Το Δεκέμβριο του 2014, για παράδειγμα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η απροσδιόριστη διάρκεια στρατιωτικής θητείας θα είναι 18 μήνες πλέον για τους καινούριους. Είναι μια σημαντική απόφαση αυτή, γιατί ήταν να προσδιορίσει τη διάρκεια της αρχαιοτικής θητείας, κάτι που ανάγκαζε πάρα πολλούς πολίτες της χώρας να μεταναστεύουν. Τώρα βέβαια μένει να εφαρμοστεί η απόφαση αυτή. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανακοφίσουμε τον πληθυσμό της Ερυθρέας και όσον αφορά την έλλειψη τροφίμων και την έλλειψη οικονομικών προοπτικών και ευκαιριών. Έχει μεγάλη σημασία το ότι ο κόσμος φεύγει, οι νέοι κυρίως, οι οποίοι ξεκινούν ένα επικίνδυνο ταξίδι προσπαθώντας να φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση παράνομα. Και γίνονται βέβαια θύματα των ε, λαθροδιακινητών. Βάσει τον Αναπτυξιακού Ταμείου, 53,7 εκατομμύρια ευρώ έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να καλύψει την περίοδο 2008 μέχρι τώρα έχει να κάνει κυρίως με την ασφάλεια ε, τροφίμων και τη γεωργία. Ο δεύτερος τομέας είναι η οικοδόμηση ικανοτήτων και η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, κυρίως μέσω των ε, κοινωτικών δικαστηρίων. Η βοήθειά μας δίνεται μέσω προγραμμάτων και όχι μέσω ενίσχυσης στον προπολογισμό. Υπάρχουν και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου προκειμένου η βοήθειά μας να φτάνει στον κόσμο απευθείας, να δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης και να μειώνεται η φτώχεια. Δεν υπάρχει στήριξη προς την κεντρική κυβέρνηση της χώρας. Όσον αφορά τώρα τον προγραμματισμό της βοήθειας βάσει του 11ου προγράμματος, οι συζητήσεις συνεχίζονται. Προβλέπεται ότι η αναπτυξιακή ευρωπαϊκή βοήθεια θα στηρίξει την κοινωνική ανάπτυξη μέσω πρόσβαση σε πηγές ενέργειας για να υπάρχουν αυτά αποτελέσματα για τον πληθυσμό. Για παράδειγμα, δημιουργία περισσότερων θέσεων απασχόλησης και βελτίωση των συνθήκων ζωής των κατοίκων εκεί. Επιπλέον, στήριξη στην ε, διακυβέρνηση δραστηριοτήτων υπέρ της ανάπτυξης. Και αυτό προβλέπεται. Πέρα από τη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης χορηγήσει και αναθέμα κονδύλια προκειμένου να στηρίξει τις ε, ικανότητες των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, τόσο των ε, κυβερνητικών όσο και των ε, μη. Παρόλο βέβαια που το πλαίσιο επιτρέπει να γνωρίζουμε ελάχιστα πράγματα, παρόλα αυτά εμείς συνεχίζουμε αυτή τη σχέση, την ενθαρρύνουμε και ενθαρρύνουμε και τη συμμετοχή των πολιτών, τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Επιτρέψτε μου να πω και δύο λόγια για τη μετανάστευση. Η Ερυθρέα είναι μια χώρα κλειδί όσον αφορά την προέλευση των μεταναστών που φτάνουν στις χώρες μας. Ο κόσμος στην Ερυθρέα θέλει να βελτιώσει τη ζωή του, γι' αυτό και η αναπτυξιακή βοήθεια θα βοηθήσει να καταπολεμηθούν οι αιτίε που οδηγούν στη μετανάστευση. Η Ερυθρέα είναι ενεργό εταίρο και στη διαδικασία του Χαρτούμ. Βάσει τη διαδικασία αυτή, τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με τους μετανάστε και τους πρόσφυγες συζητιούνται, όπως αποφασίστηκε στην Υπουργική Απόφαση του Νευρίου που μας πέρασε στη Ρώμη. Η αναπτυξιακή μας βοήθεια είναι κάτι που πρέπει να δούμε και στα πλαίσια της περιοχής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν προσπαθεί να ενισχύσει το ρόλο της Ερυθρέας. Οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ιεμένη είναι επίσης κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό και μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην σταθερότητα στην περιοχή και στην Ερυθρέα, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά δίπλα στην ε, Ερυθρά θάλασσα ο πληθυσμός πρέπει να είναι λιγότερο ευάλωτο στην ριζοσπαστικοποίηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να συνεισφέρει στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Ευχαριστώ να ακούσω τις δικές σας απόψεις για τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην Ερυθρέα και για τη συνεργασία με τη χώρα αυτή. Ευχαριστούμε κύριε Μιμιτσά. Ακολουθούν τώρα οι ομιλητές εξ των πολιτικών ομάδων. Ξεκινούμε με τον κύριο Στήρ για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η Ερυθρέα είναι μία από τις φτωχότερες χώρες στον κόσμο. Σύμφωνα και με τον δίκτυ ανάπτυξης είναι 117η μεταξύ 118 χωρών. Είναι λοιπόν σχεδόν η τελευταία χώρα έχει 6 εκατομμύρια κατοίκων, αλλά 30% των αιτήσεων για πολιτικό άσυλο προέρχονται από πολίτες της Ερυθρέας και ο λόγος είναι η κατάφορη καταπίεση και η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθρέα. Αυτό διαρκεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι έχουν ζητήσει να, οι οποίοι χαρακτηρίζουν μάλλον την Ερυθρέα, Αφρικανική Βόρεια Κορέα ή τη μεγαλύτερη ανοιχτή φυλακή του κόσμου. Τι κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο ανάπτυξης, όπως είπε ο κύριος Επίτροπος, οι προτεραιότητές μας συνδέονται άμεσα με την αγροτική ανάπτυξη και την ανάπτυξη της παραγωγής τροφίμων. Κανείς δεν αμφιβάλλει για τη σημασία που επέχει η παράδοση αυτής της βοήθειας προς τον πληθυσμό της ε, Ερυθρέας. Αλλά δεν πρέπει να φτάσει η βοήθεια αυτή στις υπηρεσίες της δικτατορίας παρά στους πραγματικούς δικαιούχους. Είναι απαραίτητο λοιπόν να έχουμε θεσμούς οι οποίοι να είναι περιεκτικοί και να συμπεριλάβουμε και τα, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο 11, 11ο πρόγραμμα για την ανάπτυξη στην Ερυθρέα. Αν θέλουμε να υπάρχει μια κοινή πολιτική εξωτερικών θεμάτων και ασφάλειας, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε την ανθρώπινη ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο έργο μας. Δεν πρέπει να τρέφουμε ψευδεστήσεις. Η πολιτική ανάπτυξης δεν μπορεί να είναι ένα υποκατάστατο της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και εξωτερικών θεμάτων. Πρέπει να εξασφαλιστεί ο σεβασμός των ανθρωπινών δικαιωμάτων στην Ερυθρέα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Στία. Για δύο λεπτά η κυρία Βαλενθίανο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι η Ερυθρέα είναι μια χώρα ξεχασμένη σε μια ήπειρο που είναι και η ίδια ξεχασμένη. Δεν ε, αναφέρεται παρά μόνο σπάνια στις συζητήσεις μας κύριε Επίτροπε δίνουμε πολύ λίγη σημασία στην Ερυθρέα και έχουμε κάνει πολύ λίγα πράγματα για την Ερυθρέα. Μια χώρα που υπάρχει υψηλός βαθμός καταστολής από τους μεγαλύτερους στον κόσμο με ένα αιμοσταγή δικτάτορα ο οποίος επί 20 χρόνια μονοπολεί όλη την εξουσία στην Ερυθρέα που είναι πια μια ανοιχτή φυλακή. <clears throat> Αλλά όταν μιλάμε για την Ερυθρέα δεν είναι μονάχα γιατί μας αφορούν και μας ε, ε, απασχολούν τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και γιατί είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των πολιτών της Ερυθρέας που φεύγουν από τη χώρα τους, προσπαθούν να βρουν άσυλο ως πρόσφυγες ή απλώς να μεταναστεύσουν σε άλλες χώρες. Αυτό μας κάνει να μιλάμε για την Ερυθρέα. Είναι μια χώρα με περιορισμένο πληθυσμό, 6 ε, εκατομμύρια, 300.000 από αυτούς εγκατέλειψαν πέρσι την χώρα τους. Πολλοί από αυτούς που εγκατέλειψαν τη χώρα τους είναι παιδιά, είναι νέοι. Οι περισσότεροι βρίσκονται τώρα σε στατόπεδα προσφύγων και αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα με τη διακίνηση των ανθρωπίνων όντων και με τα βασανιστήρια που υφίστανται στη Χερσόνησο του Σινά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να τριπλασιάσει τη βοήθεια που δίνεται μέχρι στιγμής. Αυτό είναι καλό, αλλά το θέμα είναι αν αυτή η βοήθεια θα δοθεί πράγματι στους πολίτες της Ερυθρέας ή θα υποστηρίξουμε στο status quo και την δικτατορία στην Ερυθρέα. πώ ξέρουμε ότι αυτά τα χρήματα δεν θα βοηθήσουν το δικτάτορα τη Ερυθρέα όπω έχει γίνει μέχρι τώρα. Μιλάμε για άσυλο και οικογενειακή επανένωση. Εκεί πράγματι <clears throat> αυτό είναι απαραίτητο να βοηθήσουμε του πολίτε της Ερυθρέα. Θα πρέπει εκεί να δώσουμε την έμφαση και θα πρέπει να δημιουργήσουμε και χώρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα άτομα αυτά για να μπορούν να έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση. Αυτό το οποίο δεν θέλουμε να δίνουμε την εντύπωση ότι εμείς απλώς θέλουμε να δώσουμε λεφτά για να αντιμετωπίσει κάποιος άλλος το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βαλεντιάνο, ο κύριος Χένκελ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μπορώ να προσυπογράψω όλα αυτά τα οποία ελέγχθηκαν και αυτά που είπε η κυρία Βαλεντιάνο προηγουμένως. Και πάλι αντιμετωπίζουμε τα συμπτώματα και όχι τη ρίζα του προβλήματος στην Ερυθρέα. Φυσικά έχουμε να κάνουμε με ένα διεφθαρμένο διεκτατορικό καθεστώς που δεν σέβεται τις ανθρώπινες αξίες και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και θα πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε κυρώσεις εναντίον αυτού του κράτους. Εγώ είμαι πεπισμένο ότι θα πρέπει <clears throat> να δράσουμε περισσότερο για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι καταπιέζονται <clears throat> από τη δικτατορία της Ερυθρέας. Και να βοηθήσουμε όλους αυτούς οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να φύγουν από την Ερυθρέα, αυτών που, που πρέπει να παγώσουν επίσης τα στοιχεία του, το ενεργητικό τους και αυτών που στέλνουν τα παιδιά τους σε σχολείες ελίτ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Αμερική. Αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε πια. Ευχαριστώ για δύο λεπτά. Η κυρία Μπεσέρα Μπαστερετσέα. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε Μίμητσα, η Ερυθρέα είναι μια από τις χώρες που έχει υπογράψει τη Συμφωνία του Κοτονού και όλοι όσοι έχουν υπογράψει συμφωνία αυτή λένε ότι προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από το 1993 δεν υπήρξαν εκλογε στι χωρε αυτε Πριν από ένα χρόνο ο προεδρο Αφεβέρκη είπε ότι αν αυτή η χώρα πιστεύει ότι θα έχει δημοκρατία και πολλά κόμματα, α πάει αλλού. Μιλάμε για μια κυβέρνηση που συνεχώ χρησιμοποιεί την κατάσταση έκτακτη ανάγκη. Τα παιδιά, οι γυναίκε, οι άντρε με το ζόρι πηγαίνουν να κάνουν στρατιωτική θητεία προς διόρυτης διάρκεια. Βασανίζονται, δεν υπάρχει ελευθερία έκφραση, μετακίνηση ή θρησκευτική ελευθερία και υποστηρίζουν και τρομοκρατικές ομάδες. Πρέπει νομίζω να αξιολογήσουμε τι κάνουμε με την ε, Ερυθρέα. Όμως, Σουδάν, ε, Σινάη, ο γιατρός του πηγαίνει σε όλες αυτές τις χώρες και μας εξηγεί πως οι άνθρωποι φεύγουν από εκεί για να γλιτώσουν. Και κατάφερε ο άνθρωπος αυτός να σώσει πάρα πολλούς από το Σινάη. Οι περισσότεροι είναι κάτω των 15 ετών και έχουν να διοικηθούν φοβερές ιστορίες. Όλοι αυτοί που έχουν φτάσει στην ε, Λαπετούσα ή αλλού. Λέει ο Σχαχά ότι θέλουν, ότι είναι σαν να ακούνε τις φωνές των συγγενών τους, τους οποίους βασανίζουν στη χώρα, με φοβερά βασανιστήρια. Κάποιος που σώθηκε είπε ότι πληρώνεις μέχρι και 45.000 δολάρια. Αλλιώς την έχει άσχημα. Προς το παρόν, ντάδες να ελευθερώσει οι Αφγανές. Όμως, κάποια μέρα η Ερυθρέα δεν θα πρέπει απλώς να ανήκει στην κατηγορία που μας είπε ο Πανκιμούν σήμερα το πρωί, αλλά η Ευρώπη πρέπει να βγάλει τον κόσμο από αυτή την καταπίεση, από την καταστολή, από την μη προστασία, το μη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστούμε κυρία Βασέρα Πεστερέτσε. Επόμενο ένα λεπτό κυρία Βεριζιά. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω το σύνολο των πολιτικών ομάδων που δέχτηκαν η συζήτηση αυτή επιτέλου να μπει στην ημερήσια μα διάταξη. Η διαδικασία του χαρτού μου που ξεκίνησε από την Ιταλική Προεδρία προ τι Ιταλικ... πρώην Απικίε θέλει να δημιουργήσει μία νέα κατάσταση για την Ερυθρέα. 312 εκατομμύρια ευρώ είχαν αρχικά προταθεί και μετά η πληροφορία αυτή εξυφανίστηκε από το site της Κονισιόν. Τελικά 122 εκατομμύρια τελικά, που τελικά μειώθηκαν στα 52 λόγω της μη εφαρμογής. Η Ερυθρέα είναι η δεύτερη εθνικότητα των όσων ε, διασχίζουν την Μεσόγειο για να έρθουν στην Ιταλία. Τρία σχέδια μετανάστευση χρηματοδοτούνται, ε, στη, χρηματοδοτούνται στην Ερυθρέα. Καταρχήν, αύξηση των δυνατοτήτων της κυβέρνησης Ερυθρέας να καταπολεμήσει το εμπόριο ανθρώπων. Αυτή η κυβέρνηση, κύριε Επίτροπε, μόλις δήλωσε ότι οι υπεύθυνοι και οι οργανωτές είναι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι δημοσιογράφοι της Δύσης. Πριν από δύο χρόνια ήταν η Δυσία. Με ποιον θα, συνεργα... θα συνεργαστείτε αν όχι με αυτήν την ε, διεφθαρμένη ε, κυβέρνηση και τους παρατρεχάμενους της. Ε, κινδυνεύουμε να χρηματοδοτήσουμε ένα νέο κύμα καταστολής όπου δεν μπορούμε πια καν να ξέρουμε πόσοι είναι οι φυλακισμένοι δημοσιογράφοι και που οι μισοί από αυτούς έχουν πεθάνει ε, στις φυλακές. Τώρα, το Σύνταγμα δεν έχει ποτέ εφαρμοστεί και δεν υπάρχει καν ποινικό κώδικας και εκεί με ποιον θα συνεργαστείτε. Και τέλος, ε, οι εκστατείες ευαισθητοποίησης. Τι θα χρηματοδοτήσετε και κυρίως ο Πρόεδρος Διακόπτη. Ευχαριστώ πολύ. 1,5 λεπτό η κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, η συζήτηση αυτή δεν έχει να κάνει μόνο με την Ερυθρέα μόνο. Ο Επίτροπος Μίμητσα τον Μάρτιο σε συνέντευξη τύπου αναφέρθηκε στην αναπτυξιακή βοήθεια για την Ερυθρέα και αναφέρθηκε σε ένα ποσό το οποίο μας εξέπληξε και Έκτοτε ξέρουμε πόσο πολλοί μετανάστες φεύγουν από τη χώρα. Ο Επίτροπος λοιπόν αναφέρθηκε στα σχέδια για την αναπτυξιακή βοήθεια. Κατά το παρελθόν είχαμε επίση αναπτυξιακά κονδύλια για την Ερυθρέα. Τι έγινε όμως. Τελικά δεν καταφέρουν τα χρήματα αυτά να πάνε εκεί που πρέπει, σε υποδομές, στους πολίτες, στους εργαζόμενους, τη στιγμή που αυτοί δεν κάνουν τη δουλειά καν. Ευχαριστώ, αλλά είναι κατανικαστικά έργα από πλευρά τη κυβέρνηση τους υποχρόνου, δηλαδή. Μπορώ να φανταστώ λοιπόν ότι τώρα και πάλι προσπαθούμε να στείλουμε κονδύλια, αλλά αναρωτιέμαι, ο Επίτροπος πιστεύει ότι μετά από πέντε χρόνια θα αλλάξει κάτι. Τέλος, Πρόεδρε. Όταν εμείς μιλάμε για τους αναπτυξιακούς μας στόχους και τη μετανάστευση, δεν πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε ποτέ, γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε αυτήν ε, τη βοήθεια για να έχουμε περισσότερους μετανάστες. Όχι, πρέπει τα χρήματα να πηγαίνουν στον κόσμο εκεί ώστε να μείνει στη χώρα του και να μην φεύγει. Ευχαριστούμε. James. Δύο λεπτά κύριο Τζέμις. Η κυρία Τζέμις καλύτερα. Πριν από λίγες μέρες η κυρία Νίνα Γκίλ έλαβε το λόγο στην Ολομέλεια και είπε ότι χρειάζεται εμπόριο και όχι βοήθεια ο αναπτυσσόμενος κόσμος. Και έχουμε ενωπιόν μας μια μελέτη που το καταδεικνύει αυτό απόλυτα. Η Ερυθρέα ως κράτος έχει απόλυτη έλλειψη ελευθερίας του τύπου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το 2011 η χώρα αυτή δεν επέτρεψε την είσοδο σε ένα ανεξάρτητο <clears throat> δημοσιογράφο Εθνών από φόβο του τι θα μπορούσε να βρει και η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά και πάλι αυτή τη εβδομάδα να απελευθερώσει δημοσιογράφους που κρατούνται στις φυλακές. Αλλά πλήττεται η Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο από τη δική της υποκρισία και τις ψευδεσίες της για το τι μπορεί να επιτύχει η αναπτυξιακή βοήθεια. Δίνουμε βοήθεια σε δικτάτορες και μετά θέλει να αντιμετωπίσει το κύμα μεταναστών που έχετε στην Ευρώπη. Πετάει λεφτά δεξιά και αριστερά χωρίς καμία λογοδοσία. Υπάρχουν ε, κυρώσεις οι οποίες βλάπτουν τους αθώους πολίτες και δεν αγγίζουν τους ένοχους. Η έκθεση αυτή λοιπόν ανέφερε ότι το ΑΕΠ της ε, Ερυθέας αυξήθηκε κατά 2,1% διπλάσιο από ότι το 2013. Αυτή η χώρα έχει χρυσό σίδηρο, Μικέλιο και Χαλκό. Έχει πόρους που άλλες χώρες θα ονειρευόντουσαν να έχουν στη διάθεσή τους. Αυτό το οποίο χρειάζεται η Ερυθρέα είναι να υποχρεωθεί να διαφοροποιήσει την οικονομία της, να ξεφύγει μονάχα από την εξόρυξη. Χρειάζονται θέσεις εργασίας, ασφάλεια στην εργασία τους και τη δυνατότητα να διαφύγουν την ένδια. Η αναπτυξιακή μας βοήθεια δεν αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για το πώς χρησιμοποιούμε αυτή τη βοήθεια και τι ζητούμε ως αντίτιμο από τις χώρες αυτές που δίνουμε. Και δεν νομίζω ότι ακολουθούμε τη σωστή αντιμετώπιση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τζέιμς, ο κύριος Μποργέτσιο για ένα λεπτό. Ενώ μιλάμε για κριτήρια για να αλλάξουν ε, οι, οι επιδοτήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα πρέπει να ομολογήσουμε σαφώς πως όλες οι αναπτυξικές πολιτικές προς την Αφρική είναι μια αποτυχία. Δεν είναι αποδεκτή αυτή, αυτός ο πόρος των 312 εκατομμυρίων προς την Ερυθρέα ενώ γνωρίζουμε πως δεν θα λυθεί κανένα πρόβλημα. Μάλλον θα χρηματοδοτηθεί μια λίγο διαφανής μήκυο και κυρίως η δημόσια δίκηση της διεφθαρμένης κυβέρνησης αυτής της χώρα θέλουμε σε όλα τα κοινοτικά κονδύλια τα οποία να γίνει μια αυστηρή επαλήθευση, το ίδιο να γίνει και με την ανθρωπιστική βοήθεια. Πρέπει να δούμε μια να γίνει ένας έλεγχος όσον αφορά την επίτευξη των στόχων και τη διαφάνεια των διαδικασιών. Θα πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι κινδυνεύουμε να πληρώσουμε διπλά μέσω της μαζικής μετανάστευσης, διότι επανειλημμένως ανεφέρθη ότι ένα μεγάλο τμήμα των ε, προσφύγων είναι από την Ερυθρέα. Οι αδικίες που γίνονται σε αυτή τη χώρα διακόπτει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Μποργέ. Γέζιο. Ο κύριος για δύο λεφτά. Κύριε Πρόεδρε, στο Κοινοβούλιο σήμερα Μιλάμε για αναπτυξιακή βοήθεια για την Ερυθρέα και για κατάχρηση, παραβίαση μάλλον ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το ε, καθεστώς. Εγώ θα ήθελα να θυμίσω ένα νούμερο, 5.000. Την Πέμπτη την τρίτη συγγνώμη, 2 Ιουνίου, 5.000 μέρες θα είναι από τότε που ο Ντέιβιτ Άιζακ συνελήφθη και φυλακίστηκε στην Ερυθρέα. Πρόκειται για έναν ε, Σουηδό δημοσιογράφο που βρίσκεται στη φυλακή από το 2001 υπό φρικτές συνθήκες, χωρίς καμία δίκη και χωρίς καμία επαφή με τον έξω κόσμο. Πρόεδρε, είναι μία από τις πιο σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουμε δει τουλάχιστον ε, στην Σουηδία. Πραγματικά πρέπει να ασκηθεί πίεση στη ε, δικτατορία της Ερυθρέας. Το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς έλαβαν μέτρα ώστε να σταματήσουν την την επιβολή από πλευράς των πρεσβειών της Ερυθρέας ε, επιβολής επιθέσεων κατά των πολιτών τους που ζουν στο εξωτερικό. Η Ένωση θα πρέπει εδώ να βοηθήσει γιατί θα πρέπει να πάψει η ροή χρημάτων προς τη δικτατορία της ε, Ασμάρα. Και επίση θα πρέπει να γίνει και ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Πραγματικά η Ένωση πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να σταματήσει αυτό το παράνομο καθεστώ τον τρόπο με τον οποίο ε, ε, επιβάλλουν στον κόσμο να πληρώνει για ε, επιθέσει. Θα πρέπει να επιβληθούν κυρώσει στου εκπροσώπους αυτή τη δικτωρία και όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια, που είναι το θέμα μα σήμερα, Θα το συνδέσουμε με απαιτήσει, με όρου τα ανθρώπινα δικαιώματα να εφαρμοστούν στην πράξη. 5.000 μέρες, 5.000 ε, φυλάκιση του David Isaac και οι φυλακές στην Ερυθρέα είναι γεμάτες από ένα σωρό αθώους ανθρώπους που είναι αντρισίες συνείδηση ε, και ε, στην αντιπολίτευση. Πρέπει λοιπόν να επιβάλλουμε πολύ πιο αυστηρές κυρώσεις απέναντι στο καθεστώς της Ασμάρα. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε. Και τώρα για δύο λεπτά η κυρία Κιάνγκε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από την αρχή του 2015 πάνω από 10.000 είναι οι πρόσφυγες από την Ερυθρέα που έφτασαν μόνο στις ακτές της Ιταλίας. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που φεύγουν ε, τρέχοντας από την Ερυθρέα και, και εμπιστεύονται τους ασυνείδητους ε, ε, διακινητές. Είναι δύσκολο να μιλήσουμε για αυτή τη χώρα χωρίς να δούμε το πρόσωπο των ανθρώπων που κατά χιλιάδες φτάνουν στις ακτές μας. Δυστυχώς νεκροί. Ε, εδώ και πάνω από 20 χρόνια η κυβέρνηση αυτής της χώρας ε, είναι η ίδια ομάδα. Ε, και υπάρχει μια δίθεν εναλλακτική ε, εναλλαγή μέσω δημοκρατικών δίθεν εκλογών. Ε, πολύ αίμα χύνεται στα σύνορα της Ένωσης μας και πρέπει να στηρίξουμε την ανάπτυξη αυτής της χώρας. Γι' αυτό το λόγο, κύριε Πρόεδρε, η ανθρωπιστική βοήθεια που έχει δοθεί στην Ερυθρέα εντός αυτής της προσέγγισης που επανελειμμένα έχουμε ορίσει και εδώ την προσέγγιση ότι να μπορούμε να παρέμβουμε στις, στα αίτια θα πρέπει να σπάσουν αυτή τη σιωπή. Θα πρέπει η κυβέρνηση της Ασμάρα να έρθει στο τραπέζι του διαλόγου και της ειρήνευσης, να συζητήσει χωρίς ταμπού, χωρίς να κρύβει τίποτα, ε, ενώ θα συνοδεύουμε τη χώρα αυτή σε μια διαδικασία εκδημοκρατισμού, ενώ θα στηρίζουμε τις αξίες μας και τους στόχους μας. Πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να ε, κάνουμε επαλήθευση και έλεγχο για αυτή τη βοήθεια, να εξασφαλίσουμε ότι θα φτάσει στον κόσμο και ότι θα τον ωφελήσει. Θα πρέπει να εγγυηθούμε την παρουσία και την εργασία των ανθρωπιστικών οργανώσεων στην χώρα, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των, ε, του λαού. Δεν μπορούμε να γνωρούμε, κύριε Πρόεδρε, να γνωρούμε τις συνέπειες ε, της έντασης ε, που επικρατεί ανάμεσα στην Ερυθρέα και την, την Ερυθρέα και την Αιθιοπία. Ε, θα πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη να προστατέψουμε, να προωθήσουμε την ειρήνη και το θάρρος να ξεκινήσουμε ένα διάλογο όσο γίνεται πιο σύντομα. Πρέπει να σπάσει αυτή η σιωπή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η Ευρώπη έχει αναλάβει κάποιες υποχρώσεις απέναντι στην Ερυθρέα. Μια χώρα που είναι πολύ φτωχή και οικονομικά και κοινωνικά και σε δικτατορία. Έχουμε υποχρώσεις γιατί είναι μια χώρα που έχει υποφέρει από την απεικιοκρατία και γι' αυτό έχουμε υποχρέωση απέναντί της. Ο ελεύθερος κόσμος βέβαια θέλει να καταπολεμήσει τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συγχρόνως θέλει να στηρίξει τον πληθυσμό. Ακριβώς αυτό πρέπει να κάνουμε, να στηρίξουμε τον πληθυσμό κατευθείαν εκεί. Η βοήθεια αυτή δηλαδή θα πρέπει να ελέγχεται. Συμφωνώ με την κυρία Σαρτζεντίνη η οποία είπε ότι πρέπει να ξαναδούμε την βοήθεια που δίνουμε να την αξιολογήσουμε και πάλι, γιατί δεν πρέπει να πηγαίνουν χαμένα τα χρήματά μας. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε εγρήγορση για να πετύχουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ένα λεπτό, η κυρία Σπινέλη τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πλέον σαφή ε, χάρη στο Wikileaks, οι τρόποι με τους οποίους θέλει να σταματήσει τους μετανάστες η Ευρώπη. Η χρήση βίας θα πρέπει να χρησιμοποιείται στη διάρκεια της ε, ε, επιβίβαση αλλά και όταν κατεβαίνουν στη γη. Θα πρέπει, συνεχίζουν να στηρίζουν τις ε, ελπίζοντα πω έτσι θα σταματήσουν την έξοδο. Και η πρώτη από όλου την Ερυθρέα. Ε, οι εκθέσεις οι οποίες ε, έρχονται από την Ερυθρέα είναι φρικιαστικές όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ σας παρακαλώ να ακούσετε τις εκκλήσεις των προσφύγων. διαβάζοντα ε, διαβάζοντας τέτοιες εκθέσεις, ο φυγάς θα ε, σκεφτεί πως ε, ο οποίος πρόσφυγας διαβάζοντας αυτά εδώ θα πει ότι είτε τον ε, περιορίζουμε στην έρημο της Λιβύης είτε θέλουμε να τον περιορίσουμε στα τόπεδα των προσφύγων. Δεν ξέρω πώς αισθάνεστε εσείς αλλά ξέρω πώς αισθάνονται οι πρόσφυγες. Είναι καταδικασμένοι να χτυπούν πάνω στους τοίχους που ορθώνει η Ευρώπη μπροστά τους. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό κύριε Σεμπάγιος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. ο Επίτροπος και η Σουηδοί συναδελφός μου μίλησαν για τον David Άισεχ, ο οποίο είναι δημοσιογράφος και είναι από το 2001 στη φυλακή. 5.000 μέρες στη φυλακή, σχεδόν 14 χρόνια. 13 χρόνια και 260 μέρες. Σύμφωνα με την Amnesty International, είναι ο μόνος πολίτης τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος είναι στη φυλακή αυτή τη στιγμή, λόγω των απόψεων που διατύπωσε. Υπάρχει πίεση από τη Σουηδική κυβέρνηση και υπήρξε και σιωπηρή διπλωματία. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχουν βοηθήσει για την απελευθέρωση του David Άισακ το 2009. Ο πρόεδρος Γουέκη είπε ότι δεν έχει καμία απολύτως πρόθεση να, κάνει, να οργανώσει δίκη για τον κύριο Άισακ, ούτε να τον ε, απελευθερώσει και η πίεση της Σουηδίας δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη από αυτόν. Γιατί λοιπόν δίνουμε βοήθεια. Στη Σουηδία δεν υπάρχει καμιά υποστήριξη για να δώσουμε υποστήριξη στην Ερυθρέα. Αναρωτιέμαι λοιπόν, η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση τι θα κάνει για να εξασφαλίσει ότι ένα πολίτη τη Ευρωπαϊκής Ένωση μπορεί επιτέλου να απελευθερωθεί από τη φυλακή τη Ερυθρέας. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό ο κύριος Επιτήριος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία από τις χώρες της Αφρικής με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να ενισχύσει τους δεσμούς είναι και η Ερυθρέα. Η κυβέρνηση της χώρας αυτή όμως παραβιάζει συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα η περίπτωση της ερυθρέας είναι χαρακτηριστικό δείγμα της νοοτροπίας που διακατέχει τη φιλοσοφία της εξωτερικής πολιτικής ευρωπαϊκής Ένωσης. στο όνομα σκοπιμοτήτων αλλά και ασαφών και αδιευκρινίστων και αφιλευόμενων συμφερόντων έχουμε την τάση να θέλουμε να αναβαθμίσουμε τις σχέσεις μας με χώρες οι κυβερνήσεις των οποίων δεν είναι δημοκρατικές και παραβιάζουν κατά τρόπο προκλητικό τις αρχές της δημοκρατίας η συνήθι δικαιολογία είναι ότι οι χώρε αυτέ έχουν μεγάλη στρατηγική αξία για την ευρωπαϊκή ένωση. ακόμη χειρότερα όμω θέλουμε να εντάξουμε κάποιε από τι χώρε αυτέ ενώ δεν πληρούν τα κριτήρια τη συνθήκη κοπενχάγη στην ευρωπαϊκή ένωση όπω η τουρκία τα σκόπια την αλβανία το Κωσυφοπέδιο. το μόνο που κατορθώνουμε να κάνουμε με αυτή την τακτική είναι να υποβαθμίζουμε το κύριο τη ευρωπαϊκή ενώσεω και να γινόμαστε πολιτικοί όμοιροι των κρατών αυτών. εάν θέλουμε να αναβαθμίσουμε το κύρος τη ευρωπαϊκή ενώσεω οφείλουμε να είμαστε θεματοφύλακες των αξιών και των αρχών της Ευχαριστώ πολύ κύριε Επιτήδια. Ακολουθεί για ένα λεπτό ο κύριο Φουντσουρίτσα. Χωρίς μικρόφωνο. Μικρόφωνο. Προσπαθήστε πιο πολύ λέει ο πρόεδρος. Προσπαθεί περισσότερο ο κύριο Φουντσουρίτσα. Α, μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε η Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Βοήθεια θα πρέπει να φτάσει τα άτομα τα οποία τη χρειάζονται περισσότερο. Στο φω τη κατάσταση στην Ερυθρέα, η αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ερυθρέα πρέπει να παρακολουθήσει από πολύ κοντά τη χρήση αυτή τη χρηματοδότηση. Πρέπει να συνεχίσει ο διάλογο με την κυβέρνηση τη Ερυθρέα βάσει του άρθρου 8 τη Συμφωνία τη Κοτονού για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει να υποστηρίξουμε του αγωνιστέ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνία των πολιτών. Φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έρευνα για τα θέματα αυτά δεν είχε καμία συνεργασία από την κυβέρνηση της Ερυθρέας και αυτή η Επιτροπή δεν μπόρεσε να έχει πρόσβαση στη χώρα. Όλα αυτά οδηγούν σε ανησυχίες σε σχέση με την απόφαση να τριπλαστιάσετε τη βοήθεια που δίνεται στην Ερυθρέα. Δεν υπάρχουν στοιχεία καμιάς πραγματικής αλλαγής σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα εκεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μειώσει στο μισό την βοήθεια που γίνεται μέχρι ότου η Επιτροπή η Ερευνά για την Ερυθρέα μπορέσει να έχει πρόσβαση στη χώρα αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Φροντσούλα. Για ένα λεπτό κύριο Δεμέσμακερ. Μάκερ. Σήμερα το πρωί ο Ιγδάλγος υπουργό υπεύθυνο για το άσυλο είπε στο ραδιόφωνο ότι ο αριθμό των ετούντων άσυλο από την Αιθιοπία και την Ερυθρέα διπλασιάστηκε αυτό το μήνα σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2014. Η κακή κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ο σημαντικότερο παράγοντα εξαιτία του οποίου αφήνουν τη χώρα του. και πολλοί από αυτού πεθαίνουν στη διαδρομή στη Μεσόγειο. Το Βέλγιο προσπαθεί να βοηθήσει του Ερυθρέου. Λίγοι όμω τα καταφέρουν να ξεφύγουν. Πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε αυτούς που μένουν πίσω, που δεν καταφέρνουν να φύγουν από τη χώρα τους. Όπως και να έχει το πράγμα, πρέπει να ξέρουμε ότι η χώρα βρίσκεται στην 181η θέση σύμφωνα με τον Δίκτυο των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη σε 187 χώρες. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι επίσης σε πάρα πολύ κατάσταση. Πρέπει να στηρίζουμε τους ανθρώπους, δεν πρέπει να στηρίζουμε το καθεστώς. Δεν πρέπει να απομακρυνόμαστε από τις αρχές μας. Τα ανθρώπινα δικαιώματα με την ανάπτυξη πρέπει να πηγαίνουν χέρι-χέρι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ντεμεσμάκερ και ένα λεπτό κυρία Χαουταλά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, πολύ σωστά είπατε ότι δεν βοηθάει η απομόνωση. Αλλά βέβαια το ερώτημα είναι πώς να έχουμε δεσμούς και σχέσεις με ένα καθεστώς που βάσει όλων των κριτηρίων είναι ένα από τα πιο καταπιεστικά ε, καθεστώτα στον κόσμο. Τι να κάνουμε με μια χώρα η οποία βρίσκεται όντως μαζί με την Βόρεια Κορία, ίσως και το Αφγανιστάν, στις πιο απομονωμένες ε, χώρες στον κόσμο. Πάντως, Πράγματι, πρέπει να βρούμε καινοτόμου τρόπου για να βοηθήσουμε με την αναπτυξιακή μα βοήθεια. Ένα παράδειγμα θα σα δώσω. Η... Όταν η Διεθνή Ομοσποδία για του Ανάπηρου είχε ένα πρόγραμμα να βοηθήσει του κοφού, για παράδειγμα, το είχε και για την Βόρεια Κορέα. Υπάρχει τρόπο δηλαδή να πείσουμε την κυβέρνηση σιγά σιγά ότι πρέπει να αποφεληθεί και ότι μπορεί να αποφεληθεί από τον άνοιγμα της χώρας. Και θέλω να σας ρωτήσω κάτι κύριε Επίτροπε. Έχουμε την διακυβερνητική αρχή για την ανάπτυξη και τις αφρικανικές χώρες. Η περιφερειακή συνεργασία πιστεύετε ότι μπορεί να βοηθήσει. Ευχαριστώ κύριε Χάουταλα. Για ένα λεπτό κύριο Στούχελ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Οι Ολλανδοί πληρώνουν φόρους κάθε μήνα δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Μπορείτε λοιπόν να φανταστείτε πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι όταν ακούν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει 3,5 εκατομμύρια στο καθεστώς της Ερυθρέας. Η Ερυθρέα που είναι μια χώρα η οποία βρίσκεται στη χειρότερη κατάσταση όσον αφορά τον δίκτυο ανάπτυξη, χειρότερα και από τη Βόρεια Κορέα. Πρόεδρε, Πώς νομίζετε ότι εγώ μπορώ να το εξηγήσω αυτό στους ανθρώπους στη χώρα μου. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Στίχερ. Για ένα λεπτό η κυρία Γκόμες. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθρέα είναι πραγματικά καταστροφική. Και αυτό περιλαμβάνει και το Σουηδό δημοσιογραφό που αναφέρθηκε. Υπάρχουν σημαντικές περιορίσει ελευθερίας έκφρασης και της θρησκευτική ελευθερίας. Είναι μια καθημερινή πραγματικότητα. Μετά από την ε, ανεξαρτησία του 1993 ποτέ δεν εφαρμόστηκε το Σύνταγμα. Εξακολουθεί να υπάρχει η υποχρεωτική θητεία για απεριόριστο χρονικό διάστημα, κάτι το οποίο υποχρεώνει πολλούς πολίτες Ερυθρίας να φύγουν ως πρόσφυγες και να αναζητήσουν την τύχη τους στις χώρες της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτό, με τον τριπλασιασμό της βοήθειας, θα λύσει το πρόβλημα. Θα αποτύχει παταγωδός αυτή η πολιτική, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια καταστολή στην ε, Ερυθρέα, χάρη στις ε, προσπάθειες του Πρόεδρου της δεν μπορούμε λοιπόν να διαπραγματευόμαστε με μια δικτατορία η οποία παραγνωρίζει και περιφρονεί τις δημοκρατικές αρχές που εμείς υποστηρίζουμε και με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά δρούμε τύφλα και δεν θα οδηγήσουμε σε διακόπτη ο πρόεδρος. Σε ευχαριστώ κύριε Γκόμες. Ο κύριος Παντσέρη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω πως δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει ότι η Ερυθρέα είναι το βασικό παράδειγμα όσον αφορά τις αντικειμενικές ε, ε, αντιφάσεις εντός των οποίων αναπτύσσεται η Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Πολιτική. Γιατί από τη μια πλευρά έχουμε περισσότερους πόρους για την ανάπτυξη της χώρας στην πριν απόπειρα να σταματήσουμε την έξοδο των προσφύγων και να βελτιώσουμε την κατάσταση ε, επιτόπου, ενώ τα κάνουμε όλα αυτά σε μια χώρα όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα θα παραβιάζονται διαρκώ. Δύσκολο να βγούμε από αυτήν την αντίφαση, γιατί το να μην δώσουμε πόρου θα σήμαινε ότι θα καταστήσουμε ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση για του ε, καημένου αυτού, αλλά ταυτόχρονα θα σημαίνει ότι δεν έχουμε καμία εγγύηση ότι θα φτάσουν τα χρήματα αυτά στου ανθρώπου που δυσκολεύονται. Τι να κάνουμε, νέε δεσμεύσει τη Κομισιόν και θα πρέπει αυτό να γραφτεί. Ε, καταρχήν η βοήθεια θα πρέπει να, δι... παρακολουθείται από, συγκεκριμένα, από την αντιπροσωπεία μας στην Ερυθρία και έπειτα να άμεση ε, διόρθωση του κεφαλαίου ανθρώπινα δικαιώματα. Μόνο από αυτούς τους όρους είναι αποδεκτή η πρόταση της Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Παντσέρη. Προχωρούμε τώρα μετά την εξάντληση του καταλόγου αγορητών στη διαδικασία Catch the Eye. Έχω δύο αιτήσει περισσότερες από ό,τι μου επιτρέπει ο χρόνος. Ξεκινώ με την κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να μιλήσουμε για την Ερυθρία και για όλες αυτές τις χώρες που αντιμετωπίζουν την διαφθορά, όπου ο κόσμος είναι φυλακισμένος, όπως ακούσαμε από τους εδώ συνάδελφο. Δεν μπορούμε να τους αποφύγουμε, ούτε και να τους αφήσουμε στη μοίρα τους. Και είμαστε α, μεταξύ σφύρας και άκμων. Και, άκμονος. Ε, ε, σήμερα το πρωί ακούσαμε, από έναν, ακούσαμε έναν ε, ε παπά της Αιθιοπίας. Ε, τι γίνεται και τι κάνουν εκεί, πώς αντιμετωπίζουν το Ιμπόκο Χαράμ και πώς χρειάζονται βοήθεια για να βοηθήσουν κόσμο που δεν έχουν ε, κατάλημα, ε, τροφή ούτε νερό. Επίτροπε, σωστά είπατε ότι πρέπει να τα λύσουμε αυτά τα προβλήματα γιατί αν όχι θα συνεχίσουμε να έχουμε μεταναστευτικές ροές μεγαλύτερες από αυτές που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Είναι προς το συμφέρον μας λοιπόν να τα ρυθμίσουμε αυτά τα προβλήματα επιτόπου και ακόμα και εκεί που οι πολιτικές μας αποτυγχάνουν θα πρέπει να εξακολουθούμε εξακολουθήσουμε να προσπαθούμε ε, για να βοηθήσουμε τον κόσμο αυτό που υποφέρει τόσο πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μακίνο. Ο κύριος Καπούτο έχει το λόγο. Le tensioni in Eritrea riguardano... Εντάσει στην Ερυθρέα αφορούν και την Ευρώπη άμεσα που αυτές τις εβδομάδες αντιμετωπίζει μεταναστευτικά κύματα. Μιλάμε για το μεγαλύτερο ε, ποσοστό προσφύγων που έρχεται, μεταναστών που έρχεται. Ε, μετά, δεύτερη μεγαλύτερη μεταναστευτική ροή μετά τη Συρία. Ε, άντρες, γυναίκες, παιδιά ε, και νέοι φεύγουν. Είναι πολύ δύσκολο το θέμα και τα Ηνωμένα Έθνη τονίζουν τις πολλαπλές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων η κυβέρνηση έχει χρησιμοποιήσει και τις σχέσεις με τις γειτονικές χώρες για να, για να αγνοήσει Μάλλον έχει χρησιμοποιήσει τις εντάσεις με τις γειτονικές χώρες για να δικαιολογήσει τη χρήση του στρατιωτικού, του στρατού, για να περιορίσει τις ελευθερίες και να παραβιάσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει να θέσουμε όρους για την οικονομική βοήθεια, όπω όπως τη βελτίωση της κατάστασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Ευχαριστούμε κύριε Καπούτο. Ο κύριος Μαριάς. Κύριε Πρόεδρε, η Ερυθρέα είναι πρωταθλήτρια στην Αφρική στις φυλακίσεις δημοσιογράφων. Είναι πλέον μια μεγάλη ανοιχτή φυλακή που καταπιέζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παράλληλα την περίοδο της Αραβικής Άνοιξης στην Ερυθρέα περιόρισαν την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Στη χώρα επικρατεί επί 20 ετία κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η ηγεσία της έχει γράψει τη συμφωνία του κοτονού στα παλιά της τα παπούτσια. κυριαρχούν εκεί ο υποσιτισμός η φτώχεια η βία κατά των γυναικών και οι πολίτες της φεύγουν άρον άρον και έρχονται ως πρόσφυγες στην ελλάδα και στην υπόλοιπη νότια ευρώπη. η ερυθρέα πρέπει λοιπόν να προχωρήσει σε βαθιές δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και στην οικοδόμηση του κράτους δικαίου. Πρέπει η αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πηγαίνει στο φτωχοποιημένο λαό της Ερυθρέας και όχι στους ολιγάρχες του καθεστώτος που πρέπει να αντιληφθούν ότι η ευρωπαϊκή ένωση θα σταματήσει την αναπτυξιακή βοήθεια προς την ερυθρέα εάν δεν πάψουν άμεσα να παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μαριά. Είχατε και λίγα δευτερόλεπτα ακόμα στη διάθεσή σας. Αν δεν μιλούσατε τόσο γρήγορα θα σας είχαν παρακολουθήσει και οι ο κύριος Γιάκοφτσης έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια καλή σύγκριση είναι αυτή μεταξύ της Ερυθρέας και της Βόρειας Κορέας. Είναι κράτη τα οποία δεν σέβονται καθόλου τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ξέρουμε πολύ καλά όλα αυτά τα οποία γίνονται στη χώρα αυτή. Και αυτό όμως σημαίνει να έχουμε μια συνεκτική και εξισορροπημένη πολιτική. Νομίζω ότι αυτό που είπε ο Επίτροπος Μίμητσα στις αρχικές του παρατηρήσεις που είπε ότι η ισορροπία αυτή δεν θα πρέπει να έχει το στόχο να βοηθήσει τους δικτάτορες και να, τους δώσουν, να δώσει στο δικτάτορα χρήματα αλλά να βοηθήσει σχέδια τα οποία με κάποιο τρόπο θα μπορέσουν να βοηθήσουν τον πληθυσμό για να βελτιώσει τις συνδίκες διαβίωσής του και να μείνει στη χώρα και όχι να διακινδυνεύσει τη ζωή του στην διέλευση της Μεσογείου. Θέλω λοιπόν να υποστηρίξω αυτή την πρόταση της Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Γιακόβιτς. Πετήρ. Κυρία Πετήρ, ευχαριστώ πρόεδρε. Η κατάσταση στην Ερυθρέα είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. έχει ξεπεράσει ακόμα και την Βόρεια Κορέα όσον αφορά την λογοκρισία και την καταπίεση των ελευθεριών. Δεν υπάρχει ελευθερία τύπου και δεν είναι επικίνδυνη μόνο για δημοσιογράφους η χώρα αυτή, αλλά και για τους θρησκευόμενους, εκείνοι δηλαδή που δεν ακολουθούν τις τέσσερις αναγνωρισμένες από τη χώρα θρησκείες. Ο κόσμος που ζει με φτώχεια, ζει και με το φόβο μιας στρατιωτικής θητείας χωρίς τέλος και για καταναγκαστικά έργα. Και εκδιασμούς. 4.000 ε, πολίτες κάθε μήνα φεύγουν από τη χώρα. Μια ολόκληρη ποδοσφαιρική ομάδα μάλιστα έφυγε το 2013. Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για ανάπτυξη όσο παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Προτιμούν να χάσουν τη ζωή τους φεύγοντας από τη χώρα τους οι κάτοικοι παρά να συνεχίσουν να ζουν εκεί κάτω από απάνθρωπες συνθήκες. 14.000 έφτασαν στην Ιταλία πέρυσι με σχεδίες. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να το λύσει. Ευχαριστώ κύριος Μίκελη. Έχει το λόγο. Ο Σον Κέλλη, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Πρέπει να αξιολογούμε την ανθρωπιστική βοήθεια, ιδιαίτερα εκείνη που δίνουμε σε χώρες, οι οποίες είναι διεφθαρμένες και αυταρχικές. Και νομίζω ότι η Ερυθρέα είναι ένα κλασικό τέτοιο παράδειγμα από το 1991 έχει τον ίδιο πρόεδρο, δεν έχει σύνταγμα, δεν έχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη, δεν έχει εκλογές και δεν υπάρχει ελευθερία τύπου, κάθε άλλο. Και όσον αφορά το αναπτυξιακό δίκτυο, βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση. Δίνουμε λοιπόν αναπτυξική βοήθεια σε μια τέτοια χώρα, σε ένα τέτοιο καθεστώς. Θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να βοηθούμε τους πρόσφυγες βραχυπρόθεσμα, να έχουν κάποια ποιότητα ζωής και μετά κίνητρα να δώσουμε σε χώρες όπως η Ερυθρέα. Η αναπτυξιακή βοήθεια να δίνεται εφόσον τουλάχιστον σέβονται τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Μόνο τότε. Ευχαριστώ κύριε Κέλλη. Και τέλος ο κύριο Σουάμπ για να κλείσουμε τη διαδικασία κάτι Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η Ερυθρέα για μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πραγματικό δίπλωμα. Δίλημα, συγγνώμη. Τη μια μεριά είναι ότι υπάρχουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιστολή της ε, ελευθερίας έκφρασης, όλα αυτά πρέπει να μας κάνουν να αναρωτιόμαστε αν έχει νόημα η αναπτυξιακή βοήθεια και η συνεργασία με τη χώρα αυτή. Από την άλλη μεριά υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που ζουν εκεί κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες χάρη στην ε, αναπτυξιακή βοήθεια να έχουν προοπτικές στην χώρα τους και όχι να είναι υποχρεωμένοι να πέφτουν στα χέρια των διακινητών που τους υπόσχονται να τους φέρουν στην Ευρώπη, δημιουργώντας περαιτέρω προβλήματα στην Ευρώπη. Γι' αυτό κύριε Επίτροπε πρέπει να βρούμε μια εξισορροπημένη απάντηση. Δεν μπορούμε να πούμε μονάχα ότι αυξάνουμε τον προπολογισμό της αναπτυξιακής βοήθειας. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι είναι απαραίτητο, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να αναλάβει συγκεκριμένα μέτρα για να βελτιώσει την κατάσταση. Ευχαριστώ. Κύριε Σφάμπ, <clears throat> έχει τελειώσει και η διαδικασία ΚΑΤΣΔΙ και δίνω το λόγο για να κλείσει η συζήτηση στον Επίτροπο Μιμίτσα. I agree with the concerns and... Συμφωνώ με τις ανησυχίες και τις, τις καταγγελίες κατά της δικτατορίας και της κατάχρησης παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αναφέρατε για την Ερυθρέα. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ε, το πολύ δύσκολο πλαίσιο εντός του οποίου εργαζόμαστε. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύο επιλογές. Να ακυρώσουμε τα προγράμματα βοήθειας είτε να εστιάσουμε καλύτερα την βοήθειά μας προς αυτούς που τη χρειάζονται περισσότερο. Είμαστε της άποψης ότι είναι καλύτερο, πολύ καλύτερο να εξακολουθήσουμε να έχουμε επαφές με την Ερυθρέα μέσω των διαφορετικών μας μέσων. Έπειτα ε, θα πρέπει να... Εμείς βεβαίως συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθρέα και συμφωνώ με τις προτάσεις προτάσεις ε, που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην ε, διάρκεια της εκπόνησης του Εθνικού Ενδεικτικού Προγράμματος για την Ερυθρέα υπό το 11ο ε, Ταμείο Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Βοήθειας για να βοηθήσουμε τον κόσμο και όχι την κυβέρνηση και για να αντιμετωπίσουμε τις ρίζες του προβλήματος τη μετανάστευση. Επίσης σημειώνουμε με τη δέουσα προσοχή τις προτάσεις για την καλύτερη χρήση τη περιφερειακή συνεργασία και τις σχετικές των σχετικών δυνατοτήτων καθώ και για την ένταξη σε την ε, εφαρμογή κυρώσεων κατά του καθεστώτος της Ερυθρέας. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι βασικός μας στόχος είναι να βελτιώσουμε τη διαβίωση του λαού, του πληθυσμού και να συμβάλλουμε στην, έτσι στην σταθεροποίηση της χώρας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μιμίτσα. Έχει κλείσει η συζήτηση για το θέμα αυτό. Περνάμε τώρα στο επόμενο ζήτημα που είναι η δήλωση του Συμβουλίου και της Κομισιόν σε ό,τι αφορά τις κυβερνοεπιθέσεις κατά των μέσων ενημέρωσης και τα θέματα της κυβερνοασφάλειας. Η κυρία Καλίνα Λουκασεβίκα έχει το λόγο εξ Συμβουλίου.